Θα ήθελα τώρα να σας ενημερώσω για την υπογραφή πράξεων βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Την Τετάρτη ο Πρόεδρος Συμβουλίου και εγώ θα υπογράψουμε μια δεκάδα τέτοιες νομικές πράξεις ε, βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 74 του ιστορικού κανονισμού και θα δημοσιευθούν αυτές οι νομικές πράξεις στα πρακτικά της παρούσας ε, συνόδου. Κατόπιν η κυρία Πασκάλ Γκρινή